του Ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Νόρικα Νικολάη ε, έφυγε από 7 Ιουλίου 2014, αποχώρησε από την ομάδα του ΕΛΚ και πλέον ανήκει στην ομάδα του ΑΛΔΕ. Από την ομάδα ΑΛΔΕ, ΓΚΟΕ, ΕΛΚ, ECR και EFDD ε,